δώσουμε δυνατότητες για καλύτερη επιλογή, για καλύτερες συναλλαγές στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρέντινγκ. Ολοκληρώσαμε και το θέμα αυτό. Αύριο στις 12 θα γίνει η ψηφοφορία. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση Hirsch. Συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Για τέσσερα λεπτά έχετε το λόγο... Α, η κυρία Βόλης. Η ψηφοφορία είναι Τετάρτη, λέει η κυρία Βόλης. Α, έκανα λάθο, λέει ο Πρόεδρο, Ναι, όντω την Τετάρτη και όχι αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Νόμιζα ότι αύριο ήταν Τετάρτη. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αύριο θα συζητήσουμε για την επαγγελματική κατάρτιση, τη στρατηγική 2020 και θα ψηφίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να πω από πού ξεκινήσαμε. Υπάρχει μια ανεργία των νέων, 21%. Δηλαδή ξεπερνάμε το διπλάσιο του μέσου όρου. Έχουμε επίσης μια μεγάλη ανεργία των γυναικών και προβλήματα όσον αφορά την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των ατόμων με ειδικέ ανάγκες και περιορισμένη κινητικότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βρουν μια καλύτερη θέση στον κόσμο της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια παγκόσμια οικονομία. Είναι δικό μας καθήκον να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα επαγγελματικής κατάρτισης. Και βεβαίως ξεκίνησε η συζήτηση για τη διαδικασία της Κοπενχάγης. Διαπιστώνουμε σήμερα ότι η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 θα πρέπει να συμπεριλάβει σαν κεντρικό σημείο τους νέους, οι οποίοι δεν είναι απλώς φοιτητές, και μαθητές, αλλά κάποια στιγμή μπαίνουν στην επαγγελματική ζωή και θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και ενός άλλου κράτους μέλους της Ευρώπης από αυτό το οποίο προέρχονται. Εγώ θεωρώ ότι αν κάποιος ο οποίος πραγματικά μπόρεσε σαν νέος να εργαστεί σε μια άλλη χώρα θα μπορέσει καλύτερα να ενσωματωθεί και αργότερα στην αγορά εργασίας. Το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης. Υπάρχουν σοβαρά δημογραφικά προβλήματα τα οποία μας οδηγούν σήμερα σε μια μεγαλύτερη επαγγελματική ζωή. Άρα χρειάζονται διαρκώς νέες επαγγελματικές ε, καταρτήσεις και η διαβίου κατάρτιση και επαγγελματική ε, κατάρτιση θα είναι κάτι το οποίο σαν φαινόμενο θα γενικευθεί. Οι εργαζόμενοι όλο και περισσότερο θα γνωρίζουν περιόδους επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ευελιξία στην προσφορά μας να μπορούμε να προσφέρουμε επαγγελματική κατάρτιση από κοινού και εκ παραλίλου με την επαγγελματική δραστηριότητα και την οικογενειακή ζωή. Και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στα πανεπιστήμια, στις ανώτατες σχολές και βάσει της διαδικασίας της Μπολόνια θα πρέπει να προσφέρονται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ανταλλαγές φοιτητών Κάτι που σήμερα δεν προσφέρεται αρκετά και σε μεγάλο βαθμό στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Γι' αυτό και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι από όλες τις πολιτικές ομάδες με στήριξαν και συνεργάστηκαν μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χίρς, λέει ο Πρόεδρος. Διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Παπαδοπούλου έχει το λόγο. Ω σκιώδης εισηγήτρια χαιρετίζω την έκθεση Hirsch γιατί τονίζει τη σημασία για συνεχή ικανότητα για μάθηση και εργασία, κινητικότητα και ευελιξία στο σύγχρονο και απαιτητικό διεθνές εργασιακό περιβάλλον. Είναι αλήθεια Πώ η οικονομική κρίση έφερε ανεργία και ανασφάλεια σε όλου και ειδικά στους νέους στις γυναίκες στα άτομα με αναπηρία. για να επιτευχθούν οι στόχοι τη στρατηγικής εε 2020 απαιτείται συνεχή σωστή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο στην ευρωπαϊκή ένωση όσο και στα κράτη μέλη στοχευμένε πολιτικέ και στρατηγικέ για μείωση του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο προγραμματισμό των αναγκών των ατόμων για κατάρτιση στενότερη σχέση τη προσφερόμενη εκπαίδευση με τι ανάγκε τη αγορά εργασία. είμαι βέβαιη πω το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση η διαφάνεια και η συνεργασία αλλά και η συγκρισιμότητα των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων θα στηρίξουν ακριβώ τι ανάγκε Ευχαριστώ πολύ κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Τικάου. Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάσταση είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Γι' αυτό είναι εγγύηση για το μέλλον της Ευρώπης. Διότι ο ρυθμός της ανεργίας έφτασε για τους νέους το 20% και μιλάμε για 16% εγκατάλειψη της παιδείας. Ε, εις δε την Πορτογαλία έχουμε 40% εγκατάλειψη του σχολείου. Επομένως η σοβία κατάρτιση είναι πάρα πολύ βασικό για να καταβλήσουμε την ανεργία, να λάβουμε υπόψη βέβαια στα διαδρομίες των εργαζομένων ε, γιατί έτσι θα καθοριστεί το πόσο ευαίσθητη είναι ή στην υπόθεση σοβιάς κατάρτισης θα πρέπει το κόστος να είναι εύλογο, λογικό, θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα εύκολη ό,τι καθεστώς και να διέπει οποιονδήποτε εργαζόμενο στην αγορά εργασίας ό,τι και να έχει κάνει στο παρελθόν του οπότε θα πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη ότι χρειάζεται ευελιξία του εργατικού δυναμικού και όταν αναζητούν δουλειά και όταν έρχεται η ώρα να εκπαιδευτούν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τάντσιλα. Σας ευχαριστώ. Σήμερα ε, μία από τις πιο βασικές προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσουμε είναι η ανεργία. Η ανεργία που μαστίζει τους νέους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούμε πολύ για τον ρυθμό το ποσοστό εγκατάλειψης ε, της παιδείας του σχολείου που θα έπρεπε κάτω το 10%. Όμως θα πρέπει η παιδεία να είναι πιο κοντά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η ισοδία κατάρτιση και η κατάρτιση μέσα στο χώρο εργασίας θα αποκτούν αυξανόμενη σημασία. Να αλλάξουν οι νοοτροπίες όσον αφορά την κατάρτιση και όχι μόνο όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα αλλά και όσον αφορά τους διάφορους φορείς και τα κράτη. Θα πρέπει να αρθούν όλοι οι φραγμοί εάν θέλουμε οι Ευρωπαίοι που σήμερα φοιτούν στα σχολεία να μπορούν να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το μέλλον της Ευρώπης αλλά και να πετύχει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόρουνεν είχε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Μιλάμε για την κρίση η οποία πλήττει τους νέους, αλλά είναι μια γενικότερη οικονομική κρίση με τεράστια ποσοστά ανεργίας των νέων. Οι νέοι μας σήμερα εγκαταλείπουν την Ευρώπη και αυτό είναι μια πραγματική απειλή για την οικονομία της Ευρώπης και τη συνοχή της κοινωνίας μας τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε με την επαγγελματική κατάρτιση έτσι ώστε να γίνει η Ευρώπη πάλι ανταγωνιστική. Χρειαζόμαστε εργαζόμενους οι οποίοι πραγματικά να μπορούν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν να τους προσφέρουμε δεξιότητες, και προσόντα τα οποία είναι κάτι που θα οδηγήσουν σε μια ποιοτική προσφορά επαγγελματικών δυνατοτήτων κατάρτισης και θα πρέπει παραδείγματος χάρη να εμπνευστούμε από τα μοντέλα όπως το γερμανικό και το δανέζικο στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόγουνεν. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Κασριάη και τελειώνοντας θα δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Χίρς. Πολύ επικοδομητική προσέγγιση που ακολούθησε και θα ήθελα να πω ότι την άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον διότι ήταν δικό μου χαρτοφυλάκιο προ 12 ετίας. Ξεκίνησα προσπαθώντας να προωθήσω την κινητικότητα στην κατάρτιση, κάτι που δεν ήταν στο πρόγραμμα τότε και χαίρομαι που ακούω πόσο στεναρή η θέση του Κοινοβουλίου προσπαθώντας να αναπτύξει αυτό το βασικό στοιχείο για τη στρατηγική της Ευρώπης του 2020. Θα ήθελα να πω επίσης πόσο καλωσορίζουμε την έκθεση που ενισχύει και συμπληρώνει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου 2010. Αυτή η ανακοίνωση τροφοδότησε την αναθεώρηση της διαδικασίας της Κοπενχάγης και την, ε, η ανακοίνωση της Μπρίζ έγινε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Επαγγελματική Κατάρτιση για την περίοδο 2011-2020. Πολλές από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου ανταποκρίνονται στις προτάσεις της ανακοινώσεως της μπριους και συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να ξυγχρονίσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη, να γίνει ελκυστική να έχουμε ειδικευμένους εκπαιδευτές και διδασκάλους, καινοτόμε μεθόδους μαθήσεως, ε, καινοτόμε υποδομές και μέσα και χρειάζεται και κινητικότητα. Ε, να δώσουμε κίνητρα στους νέους και στους λιγότερο νέους να θέλουν να βγουν από το κάτω μέλος τους για να αποκτήσουν εμπειρίες. Είναι σημαντικές οι εμπειρίες. Αν θέλουμε να έχουμε πραγματική ευρωπαϊκή παιδεία και κατάρτιση και σχετικό χώρο. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πετύχει ισορροπία μεταξύ των φύλων, να βοηθήσει μειονεκτούσε ομάδες μέσω του προγράμματος διαβίου εκμάθησης, κυρίως μέσω του προγράμματος Λεωνάρδο Νταβίντσι που συμπεριλαμβάνεται. Όλη η βοήθεια του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ κυρία Ρέντινγκ. Τελειώσαμε με το θέμα αυτό και η ψηφοφορία θα γίνει πραγματικά αύριο αυτή τη φορά. Η συνεδρίαση διακόπτεται. Αύριο θα συνεδριάσουμε τις 9 στις 1.